Ja, liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, ας καθίσουμε. Για να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τις ψηφοφορίες μας. Ξεκινάμε. Στο σημείο 7 της ημερήσια διάταξης. Παρακαλώ, όσοι θέλουν να συζητάνε, να βγουν έξω από την αίθουσα. Όποιος θέλει να ψηφίσει, να μείνει εδώ. Ο εισηγητής παρακαλώ να λάβει το λόγο εάν θέλει. Θέλετε κάποια, κάποια εξήγηση τελευταία στιγμή, κάποια διευκρίνηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το ότι βγήκαν από τα άνετα περιθώρια που υπήρχαν, το comfort zone που λέμε πολλές φορές και έτσι καταλήξαμε σε βρήματα και σε συμφωνίες ε, όπως σήμερα το πρωί μεταξύ πέντε ομάδων σε αυτήν την Επιτροπή. Ήταν πολύ θεραλή απόφαση εκ μέρου όλων των ομάδων και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πάντες. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι ερχόμαστε εδώ και βρίσκουμε κοινό τόπο και προτείνουμε κάτι τέτοιο για τις κοινωνίες μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους πάντες για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ Κρίτσον. Μια μικρή αλλαγή λοιπόν, γιατί κάποιε ομάδε έχουν συμφωνήσει με την ε, συμβαστική τροπολογία. Ίσως να μην ισχύει 100% αυτό που θα έχετε στους καταλόγους των ψηφοφοριών, επομένως θέλει λίγο προσοχή. Ξεκινούμε με, τη συμβαστική, με την ενοποιημένη συγγνώμη consolidated υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 141 έχει αποσυρθεί και πάμε στην ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ας πάμε γρήγορα πιο μπρος. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Κυρία Σνέρχαρτ. Κύριος Σνέρχαρτ, ναι. Ναι, πολύ σύντομα και εγώ έχω καταθέσει εδώ τροπολογίες που έχουν μπει στην υπαριθμόν 1, έχουν υπαχθεί στην υπαριθμόν 1, αλλά αντίκειται, αλλά αντίκειται σε αυτό που θέλαμε. Γι' αυτό λοιπόν να γίνει χωριστά τα ψηφοφορία. Σε τμήματα δηλαδή, γιατί δεν αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο εγώ ήθελα, επεδίωκα με την τροπολογία μου. Μάλιστα, ο πρόεδρος. Ένα λεπτό όμως, η, το ΕΛΚ έχει συνυπογράψει την ενοποιημένη τροπολογία. Τώρα μας λέτε ότι η τροπολογία σας δεν έχει θέση εδώ. Μήπως πρέπει να τα βρίσκετε μεταξύ σας στην ομάδα εργασίας του ΕΛΚ. Από εδώ και μπρος, πώς θα χειρίζεστε τα θέματα των τροπολογιών. Καλώς. Ενοποιημένη λοιπόν τροπολογία Λοιπόν, τρία υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Κάνουμε ένα άλμα. Και εγώ, τουλάχιστον λέει ο πρόεδρος, πάω στη σελίδα 11. Με την ενοποιημένη τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και η 4. Το χωρούμε τώρα στην ψηφοφορία της τροπολογίας 23 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 24 υπέρ. Επαληθεύουμε την 23 λέει ο πρόεδρος. Επαλήθευση την 23. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Οι πράσινοι έχουν μία ψήφο περισσευούμενη. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 18 υπέρ. 23 κατά. Απορρίπτεται. 24 τώρα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ Κατά. Αποχές απερίφθη. Ενοποιημένη τροπολογία υπερθυμών 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάλι με ένα άλμα πάμε στη σελίδα 16 και την ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άλλο ένα άλμα. Στη σελίδα 18, λέει ο πρόεδρος. Όχι. Δεν είναι 18 γιατί έχει καλυφθεί. Πάμε στη σελίδα 20. Και την ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 7 την ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται άλλο ένα άλμα στην ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε στην ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «321 τώρα, τροπολογία υπαριθμών 300, 314 διότι ο 314, μια διόρθωση και ψηφίζουμε την 314 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν και ψηφίζουμε την 321. 321 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απερίφθη διορθώνει ο πρόεδρος. 322. Ψηφίζουμε την 322 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Να επαληθεύσουμε εφόσον το θέλετε. 323 ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 17 υπέρ. 31 κατά απερίφθη. Η 70 τώρα, τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ογδόντα ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο ταυτόσιμε στη συνέχεια καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία παριθμών 1 υπέρ παρακαλώ τροπολογία 1 κατά εγκρίνεται πιστεύω αλλά ας επαληθέψουμε για άλλη μια φορά Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 38 υπέρ. 13 κατά. Σαφώ έχει εγκριθεί. Οι 82 και 83 είναι ταυτόσιμε, τι ψηφίζουμε υπέρ. Κάτα. Αποχέ συγκρίνονται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 85 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε όμως ας επαληθεύσουμε παρακαλώ μια φορά ακόμα εψήφισαν όλοι πέρασε τις προφορίες. 29 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται Στη σελίδα 32 υπαριθμόν 100 τώρα, υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 101 υπέρ. εποχές συγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές Υπαριθμόν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 111 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπερθών 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε όμως. Υπαριθμόν 5, τροπολογία 5, ηλεκτρονική επαληθεύση. Εψήφισαν όλοι. Η φιλελεύθερη, η Άλντα, έχει μία ψήφο περισεβούμενη στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να βγει μία κάρτα από τα μηχανήματα. Τώρα ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. 46 πέρα 9 κατά. Προφανώς έχει εγκριθεί. Στη συνέχεια έχω την 112 και 5 της Επιτροπής Γεωργίας που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε την 112 και 5 της Επιτροπής Γεωργίας ηλεκτρονικά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα από εδώ που κάθομαι. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. 31 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση γιατί δεν είδα οι φιλελεύθεροι τι έκαναν. Εψήφισαν οι πάντες, πέρας φορέα. 22 υπέρ, 32 κατά, περίπτωση. Υπαριθμών 10 ενοποιημένη τροπολογία τώρα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 100. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει και έτσι πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ως ήθιστε άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν οι πάντες πέρα της ψηφοφορίες, 44 υπέρ. 8 κατά 3 αποχές. Και τελική ψηφοφορία για την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Και ψήφισαν όλοι. Πέρας. 36 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή και συγχαρητήρια στον Τρίτονα, Αρσένη ο οποίος σήμερα το απόγευμα με τη διάθεση για συμβιβασμό με τους σκιώδεις ηγητές μας διευκόλυνε σημαντικά. Μόλις 15 λεπτά χρειάστηκαν για όλες αυτές τις ψηφοφορίες. Αυτό το φίλουμε σε εσά κυρία Αρσένη για την πολύ καλή συνεργασία. Σε ευχαριστούμε θερμά Κρήτονα. Και πάω στην επόμενη έκθεση του κυρίου Ζιλ Παρνιού. Τροπολογία παριθμών 11 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. 51 ένα υπέρ κατά. Δεν είναι ορατό το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να επαληθεύσουμε την 51 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 57 υπέρ. Ουδεμία ψήφος κατά, καμία αποχή, προφανώς. Πέρασα. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθης, ερωποιημένη υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τώρα πάμε στην 57 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 59 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 60 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ 63 κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 λέει ο πρόεδρος. Κατά. Αποχές. απερίφθη. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 74 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 85 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 86 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη δύο ταυτόσιμες τροπολογίες 23 και 91. Θα ψηφίσουμε από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνονται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 95 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Πάλι ταυτόσημες. 97-98 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτονται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 100 υπέρ. Κατά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 105 και 106 από κοινού είναι ταυτόσιμο το περιεχόμενο υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτονται 28 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά από και σαν κρίνεται 107 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ευαληθεύσουμε. 114 ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει μία ψήφο παραπανήσει. Εντάξει, λοιπόν, 38 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται η 114. 116 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθει. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφθη. 31 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118-119 ταυτόσιμες τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά απορρίφθησαν 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. λογική σκέψη. υπαριθμό στην 33 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Υπάρχει 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική περιθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 5 τροπολογία υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 40. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. και εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. σε απερίφθη. 42 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία εψήφισαν όλοι Πέρας. 52 υπέρ. 7 αποχές. Και ψηφίζουμε πάλι ηλεκτρονικά την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι. Το ΕΡΚ έχει μια περισσευούμενη ψήφο. 52 υπέρ. 6 κατά εποχές, συγγνώμη, και συγχαρητήρια στον κύριο Πάνιο. Και συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκθέσεως στην Επιτροπή. Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Έκθεση Ρόσπαχ. Μία και μόνο ψηφοφορία. Τελική. Άρχεται η ψηφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Έγκρινεται ομόφωνα και συγχαρητήρια στην κυρία Ρόσενμπαχ. Και περνάμε τώρα Α, όχι, δεν είχαμε προβλέψει ψηφοφορία του σημείου 10, γιατί αναβάλλεται για διάφορους λόγους από τις ομάδες που το έχουν ζητήσει η ψηφοφορία αυτή και η Επιτροπή Αλίας έχει δώσει αναβολή στη δική της ψηφοφορία, άρα έχουμε χρόνο και ενδεχομένω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ λύσεις. Άρα δεν γίνεται ψηφοφορία για το σημείο 10 σήμερα και έτσι περνάω στην έκθεση Jordan. Και τώρα πάμε στο σημείο 11. χάρτη πορεία για το 2050. Η κυρία Γιόρντον με μια τροπολογία τη τελευταία στιγμής που μα την έχει μοιράσει όμω νομίζω εγκαίρω σε όλε τι ομάδε, και άρα μπορεί να γίνει η ψηφοφορία εάν μου δώσει κανεί τον κατάλογο των ψηφοφοριών λέει ο πρόεδρος. Zum konsolidierten 1. Wer ist dafür? Ενοποιημένη παρακαλώ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. παρακαλώ υπέρ κατά Wir stimmen nochmal ab mit Handaufzeigen, bevor wir elektronisch abstimmen. Wir stimmen ab über. Ψηφίζουμε την υπαριθμόν 9, παρακαλώ. Η υπαριθμόν 9 τροπολογία υπέρ, κατά, Αποχέ. η 11. Αποχέ απερίφθη. Ε, ενοποιημένη υπαριθμόν 2, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Υπαριθμόν 20 τώρα τροπολογία. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ενοποιημένη 6. επαληθεύουμε αυτό ζητάτε. Επαληθεύουμε την 20. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 31 υπέρ, 31 κατά. Και ω εκ τούτου, για μία ψήφο δίφορα, απερίφθη. Πάμε στην ενοποιημένη παριθμόν 6. Με τροποποιημένη διατύπωση, όπως σας δυναμήθηκε σήμερα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. επαληθεύσουμε για την τροπολογία αυτή ηλεκτρονικά, την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την 23 από ό,τι μου λένε ως προσθήκη. 23 ως προσθήκη, άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ την έχω σελίδα 5 του καταλόγου ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Η τροπολογία 5. Η τροπολογία 23, λέει ο Πρόεδρος, παραλαμβάνω. Ψηφίζουμε την 23 ως προσθήκη. Τροπολογία 23, σελίδα 5, ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 τώρα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίσουμε την 38 ηλεκτρονικά παρακαλώ έρχεται η ψηφοφορία 38 ηλεκτρονικός έλεγχος ψήφισαν όλοι πέρας 29 υπέρ 30 κατά απερίφθη 41. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Το δεύτερο τμήμα της 41. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 37 υπέρ, 23 κατά, 2 εποχές, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα και έτσι προχωρώ. 43 παρακαλώ, υπέρ. Άρχεται την ψηφοφορία, συγγνώμη, η ηλεκτρονική. 43 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Όχι, με, διαχειρός, Την 43 διαχειρός υπέρ. Όχι ηλεκτρονικά. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Δεύτερο τμήμα. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 44. Πάλι δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. 44 ηλεκτρονικά παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας παριθμών 44. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 33 υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 44 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Ε, εγκρίνεται διορθώνει ο πρόεδρος. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές επερίφθη 57 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε 47 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. ...32 υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη παριθμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65, στο δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα της 65, ψηφίζουμε παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά την 66 στο δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα της 66 ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 33 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. 72 δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά Άποχες. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Το ΕΛΚ έχει μία περίσσια ψήφο. Πάλι, ακόμα, ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. 52 υπέρ. 9 ψήφι κατά, 2 έχεις. Και συγχαρητήρια στην κυρία Γιόρνταν. Gut, wir kommen jetzt zum Bericht Antonescu und Αντωνέσκου. Και πάλι παρακαλώ να συγκεντρωθούμε στη συνψηφοφορία. 26, πρώτη τροπολογία, υπέρ. Τρία τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στο δεύτερο τμήμα της υπαριθμών 26 τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 υπέρ 30. Κατά απερίφθη. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απέρφεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 36 έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί, 41 τώρα, υπέρ. 42, 42 λέει ο πρόεδρος, υπέρ. Την τροπολογία 42, διότι όλες οι ενδιάμεσες η 36 έχει αποσυρθεί, η 37, 38, 39 έχουν περάσει όλες, έχουν αποσυρθεί, η 42. Βλέπω άλλωστε να συγκατανεύουν οι συνάδελφοι. Ψηφίζουμε την 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. 42 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 32 υπέρ, 31 κατά εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ. Κατά Αποχές. Απερίφθη. Σε τμήματα η 51 το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Αποχές και επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα της 51 ηλεκτρονικά. Μία ψήφος περισσεύει από το ΕΛΚ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 43 υπέρ. 20 κατά. Και έτσι εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. 54 ε, νομι υπέρ. Κατά. Αποχές επερίφθη. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρολογική επαλήθευση για την 59. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 31 ψηφί, υπέρ, 33 κατά. Απερίφθη. Τροπολογία 60. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Τρία τμήματα διόρθωνε ο πρόεδρος. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 61 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 19 υπέρ, κατά, αποχές Δεν είμαστε σίγουροι. Ηλεκτρονική επαλήθευση για 19. Ηλεκτρονική επαλήθευση, εψήφισαν όλοι. Το ΕΛΚ πάλι έχει μια ψήφο, μια ψήφο παραπανήσια, παρακαλώ, κάντε κάτι γι' αυτό. Εντάξει. 28 υπέρ, 33 κατά, απερίφθη. Και τώρα. Πάμε στην συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Μπερδεύτηκα, λέει ο πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα. τη 22 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απερίφθη. Η 23. Πάλι δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. κατά. Αποχές απερίφθη το δεύτερο τμήμα. Επαληθεύουμε το 23 δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική επαληθεύση παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, 32 κατά. Απερίφθη. 24 υπέρ κατά. Αποχές απορρεύτη 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη και κάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 57 υπέρ. Δύο αποχές. Και συγχαρητήρια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 Σημείο 13. Ψηφοφορία. Έκθεση Ροντρίγε. Ο οποίο έχει στήσει το λόγο. Εισαγωγικά για μια εξήγηση για μια δήλωση μάλλον, γιατί υπάρχει, έχει παρισχύσει κάποια αλλαγή εντωμεταξύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα λεφτάκι μόνο για να σας πω ότι όπως είπα σε κάποια φάση ότι δεν ήθελα να δώσω ολόκληρη μάχη για την τροπολογία παραθμών 1 εκεί που αναφερόμαστε σε κανονισμό, οδηγία κλπ. Έχουμε βέβαια τις κυρίες για να κουδάκι την τροπολογία. Εγώ απέσα τη δική μου όμως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ε, ότι στο 24 εκεί που αναφέρεται στα της νύχτας εκεί λέει ότι έχουμε εδώ πέρα ε, ε, μία αντίφαση. Έχουμε δύο θέσεις που αντιφάσουν μεταξύ τους. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει κανένας λειτουργικός περιορισμός όσον αφορά τις πτήσεις. Και να έχουμε full time λειτουργία το βράδυ, πλήρη λειτουργία. αλλιώς προσοχή, τέτοια κινδυνεύουμε να, να κόψουν όλες τις πτήσεις σε αντίθετη περίπτωση. Άρα αυτή εδώ η τροπολογία δεν, δεν λέει τίποτα. Γιατί αφορά όλη την Ευρώπη τον, τον, τον, τον, τον Ευρωπαϊκό Φορέα. Επομένως, εδώ υπάρχει λόγος υποβολής αυτής της τροπολογίας και αυτής της ρύθμισης. Όμως είναι ανόητο να κάνουμε μια τροπολογία προσπαθώντας να, να, να, να συμβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Την αποσύρω τη δική μου, αλλά νομίζω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική. Γιατί σας είχα πει ότι εδώ πέρα υπάρχει αντίφαση και εντάξει να την αποσύρω. Όμως με τίποτα να μην ε, καταλήξουμε να πούμε ότι δεν θα έχει νυχτερές πτήσεις. Γιατί έχουμε ένα σωρό πακέτα τα οποία υπάρχουν πτήσεις νυχτερινές και στην Κολονή παντού στην Ευρώπη. Να μην υπάρχει περισμός επομένως ε, και να υπάρχουν ε, νυχτερινές πτήσεις. Επομένως, υπήρχε εδώ πέρα καλή πρόθεση, αλλά τελικά καταλήξαμε να προτείνουμε κάτι ανόητο και υπάρχει αυτή εδώ η αντίφαση. Οπότε παρακαλώ να λάβουν τι ευχαριστίε μου επίση και γραμματεία αλλά και σκιωδησηγητέ γιατί με διευκόλυναν πάρα πολύ στη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Τον εισηγητή δεν είναι και εύκολο το θέμα που έχουμε να ψηφίσουμε. Ας πάρουμε μπρο. Η πρώτη τροπολογία είναι 51. 51 υπέρ παρακαλώ. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 63 ηλεκτρονική επαληθεύση. Περισσεύει μια ψήφος από το ΕΛΚΑ. Εντάξει τώρα. 60 υπέρ. Καμία ψήφος μηδέν. Ε, κατά. Καμία ψήφος αποχής. Και συγχαρητήρια στους συνταδέλφους για την ομοψυχία. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 65 και ψηφίζουμε την 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά επαληθεύουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 37 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67-68 μαζί υπέρ αποχές συγκρίνεται. 71 επαληθεύουμε τις 67-68 ηλεκτρονική επαλήθευση ε, ψήφισαν όλοι 29 κατά, απερίφθη. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Η 19 από ό,τι γνωρίζουμε έχει αποσυρθεί. Και ψηφίζουμε την 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχή και εποχές Αλλά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Το ΕΛΚ έχει μια ψήφο περισσεύομενη. 35 πέντε υπέρ. 26 κατά, κατά. Εγκρίνεται. 77 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθη. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 22 τώρα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την 81. 81 ηλεκτρονική επαληθεύση. Εψήφισαν όλοι. Και το ΕΛΚ ακόμα ψήφισε σωστούς αριθμούς, πέρασε προφορίες. 29 υπέρ, 30 κατά. Με ναι. Έλαξε διαφορά. Απερίφθη. 82 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 πρώτο τμήμα, αφού το δεύτερο έχει καταπέσει, λόγω της απόσυρσης της 19. Πρώτο τμήμα της 24, παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 86 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. 86 ψηφίζουμε. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 31 ψήφι κατά. Απερίφθη. 87 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απειρήφθη. 90 και ε, 91. Ταυτόσιμες. Τι ψηφίζουμε μαζί λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 26 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Ε, 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 98 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Επαληθεύουμε την 98, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 30 υπέρ. 31 ψήφι κατά. Απερίφθη. Ενενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 101. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απόχες περίφη, Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 102, αλλά μόνο το δεύτερο τμήμα της 102. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες, απερίφθη. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. 103, επαλήθευσε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. 29 υπέρ. 32 κατά. Και έτσι περίπτωση. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 28 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 110 υπέρ. Κατά. Εκατόν δέκα επαναλαμβάνω υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίσουμε το 109. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, 30 κατά. Απερίφθη. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 36 υπέρ. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37-38 μαζί. Υπέρ. εγκρινούνται. Επαληθεύουμε. 37-38 ηλεκτρονική επαληθέσεις. Πέρας της ψηφοφορίας η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ. 37 κατά. Απερίφθη. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 39 υπέρ.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 Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48-49 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 και 128 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ. Κατά. Προσπαθώ να μετρήσω χέρια, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. 123 ηλεκτρονική επαληθεύση. Ηλεκτρονική επαληθεύση. Ψήφισαν όλοι πέρας 36 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Είναι υπέρ, κατά, αποχές και ε, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 125, ποιοι είναι υπέρ, πίνε κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχή συγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε στι ιτουλικές παραγράφου και πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 52 υπέρ κατά συγκρίνεται. Υπαριθμών 2 πίνε υπέρ, είναι κατά, αποχές συγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχέ, συγκρίνεται. 4 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται 55. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 7 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 8 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 57 γιατί είναι ταυτόσιμες. Από κοινού υπέρ κατά αποχές συγκρίνονται. 56 υπέρ κατά αποχές συγκρίνονται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. είναι ναι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 καταπίπτει 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και όταν κάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. ψήφισαν όλοι. πέρα 54 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μπράβο σας. Oh, και τώρα πάμε στο σημείο 14 και 15 μαζί. Κύριε Μαγκελόν. Θα ήθελα απλά να διευκρινίσουμε και τα σημεία 19 και 20 θα εξετάσουμε σήμερα ή αύριο το απόγευμα. Μας είπαν χθε ότι αν τελειώνει η το απογευμα μας ειπαν χθε νωρίς Μπορεί να εξετάσουμε τα σημεία 19 και 20 σήμερα το απόγευμα, απλά για να είναι πιο σαφέ για του συναδέλφου. Συγγνώμη. Όχι 19, 20, 20 και 21. Ο λοιπόν, να τα ξαναπώ για να είναι σαφή για όλα, για όλους. Πρώτα απ' όλα, ασχολούμαστε με τα ζώα. Με την κυρία Σνέλχαρτ, λέει ο πρόεδρος και θα προλάβουμε πιστεύω να κάνουμε και το 21 αλλά δεν ξέρω εάν είναι εδώ κάποιος από την Επιτροπή γιατί φαντάζομαι ότι θα περιμένανε να δούμε το θέμα αυτό αργότερα. Λοιπόν, το 20 και 21 σήμερα τα κοιτάμε, τα εξετάζουμε. Η κυρία Σνέλχαρτ λέει ο πρόεδρος. Τα σημεία 14 και 15. Παρακαλώ. Ο κύριος Σνελχάρ, του πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για την πολύ συνεργασία που ενίσχυσε σημαντικά την έκθεση. Είναι σημαντική όμως συζήτηση, διότι υπάρχουν διαφορετικές βάσεις θέματα ουσίας πρέπει να ε, συζητήσουμε. Η πρώτη βασική αρχή είναι ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζεται έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την μετακίνηση μη εμπορικού χαρακτήρα ζώων πέραν των συνόρων. Άρα δεν ισχύει ο κανονισμός μέσα σε μια χώρα, αλλά μόνο σε περίπτωση διάβασης των συνόρων. Επίσης, Θέλω να υπογραμμίσω, υπάρχουν και πολλές πρωτοβουλίες εξάλλου, που έχουν να κάνουν με τα αδέσποτα. Και θέλω να υπογράψω ότι πρόκειται βέβαια για ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, οφείλουμε να επιλύσουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Θα παραπέμψω στην στρατηγική, στο έγγραφο στρατηγικής για την ευημερία των ζώων, όπου στο σήμερα 17 αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει έκθεση για τα δέσποτα ζώα που θα προτείνει ε, λύσεις βιώσιμες, διαρκείς ε, και κατάλληλες για τα κράτη-μέλη με ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των μικρών ζώων για την ε, κατάρτιση ενός μητρώου. Αυτή είναι μια πτυχή λοιπόν που απασχολεί πολλούς συναδέλφους εδώ. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε με μια μόνο κοντιλιά μέσα στη δική μου έκθεση, η οποία, όπως είπα, ασχολείται μόνο με την διασυνοριακή διακίνηση ζώων, μετακίνηση ζώων, να το επιλύσουμε. Και είναι, πιστεύω, σημαντική η διαπίστωση, την οποία εγώ τουλάχιστον κατά την επεξεργασία του φακέλου αυτό είδα συχνά, ότι εδώ πρέπει να προχωρήσουμε με το θέμα των αδεσποτών ζώων σε μια υποχρεωτική καταγραφή ε, που δεν είναι δυνατόν να επιληθεί με το σύστημα που συζητούμε εδώ. Γιατί του ή άλλως τα αδέσποτα θα μπορούν να καταγραφούν σε μια βάση δεδομένων, θα μπορούν να ε, αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικά και ότι θα μπορούν να, δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημά τους. Και εγώ θα πρότεινα το εξή. Γιατί ούτε για τα βοηθή, ούτε για τους χείρους, ούτε και για τον άνθρωπο δεν έχουμε μία ε, βάση δεδομένων εγκεκριμένη που να μας καλύπτει όλους, να μας περιλαμβάνει όλους. Δεν υπάρχει τέτοια λύση. Άρα λοιπόν το να υποχρεώσουμε την καταγραφή ιουδήποτε σκύλου και γάτας που κυκλοφορεί αδέσποτος στου δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μια ε, βάση δεδομένων είναι νομίζω πολύ υπερβολικό ως προς ε, τη δυνατότητα που έχει το δημοκρατικό μας σύστημα να επεξεργαστεί στοιχεία. Και θα είναι βέβαια και δύσκολο πρέπει να πω. Το να πούμε στην κάθε γιαγιά πήγαινε να δηλώσει τη γάτα σου. Θα μου πει τι, τι να δηλώσω. Τι να δηλώσω εμένα κάθε στον καναπέ μου. Δεν βγαίνει από το σπίτι θα πάει. Επομένω, το να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο θα θεωρηθεί και υπερβολικά αυταρχικό, για να το πω έτσι. Γι' αυτό παρακαλώ του αδέλφους όλους στην υπόθεση αυτή να επικεντρωθούμε, όπω είπα, στα ζώα που αφορά η έκθεση, δηλαδή τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων ή το εμπόριο και οι εισαγωγές και να μην ασχοληθούμε με τα αδέσποτα, διότι και κόστο και γραφειοκρατία εισάγουμε και μην ξεχνάμε ότι και το κόστος είναι σημαντικός παράγον. Και βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί είναι αυτοί που θα θέλανε να λύσουν τα προβλήματα με νομοθετικές παρεμβάσεις. Αλλά θα έλεγα, χωρίς να λησμονήσουμε το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, να μην το αντιμετωπίσουμε εδώ στο πλαίσιο της δικής μου έκθεσης, των δικών μου εκθέσεων, αλλά να το δούμε χωριστά σε μια άλλη έκθεση. Υπάρχουν τώρα διάφορες επιμέρους ε, τροπολογίες, οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Εν συντομία, η εγκατάσταση ενός ε, αναμεταδότη, transponder, από τον κτηνίατρο που προτείνεται, ε, με καταχώρηση στη συνέχεια σε ένα μητρό κτλ. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν διαφορετικές μεθόδους. Και ως εκ τούτου και εγώ λαμβάνω υπόψη το δεδομένο αυτό στην ε, σχετική μου τροπολογία. λέγοντας ότι δεν θέλω να ανατρέψω τα εσκεμένα, εσκαμένα σε ορισμένα κράτη-μέλη εφόσον ισχύουν κάποιες λύσεις αποτελεσματικά, αλλά εκείνα τα οποία δεν έχουν άλλη λύση ας εισαγάγουν τον ε, με μια μικρή παρέκκληση τώρα. Γιατί άλλο έλεγε κτηνίατρο, άλλο έλεγε δεν πειράζει χωρί κτηνίατρο. Εν περιπτώσει, εμεί λέμε να γίνει αυτή η καταγραφή και μέσω του κτηνιάτρου οπωσδήποτε, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σαφέ για να μπορεί να περάσει και τα διάφορα στοιχεία στην ταυτότητα του ζώου. Επίση, πολλέ είναι τροπολογίε οι οποίε εισάγουν ε, εξαιρέσει για τα νεαρά ζώα, πράγμα το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι πολύ καλά. Να επαναλάβω. Είχαμε πει ότι η ανοσία περνά από τη μητέρα στο νεογνώ, τις πρώτες 12 εβδομάδες δεν γίνεται εμβολιασμό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η ιατρική εικόνα του ζώου. Αλλά εάν λέει ο κτηνίατρος ότι το ζώο δεν είχε επαφή άλλη εκτός από τη μητέρα, μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται εμβολιασμό. Αλλά μένει ένα κενό δικαίου για τις περιπτώσεις από 12 έως 18 εβδομάδες. Γιατί εάν γίνει ο εμβολιασμός στις 12 ακριβώ εβδομάδε μέχρι τι 18 δεν υπάρχει απόδειξη για το αν έχει πράγματι γίνει ο εμβολιασμός. δεν βλέπουμε αντισώματα. Και άρα πάλι λέμε ότι χωρεί βεβαίωση, ότι δεν υπήρχε επαφή με άλλα ζώα, ότι η μητέρα έχει ήδη εμβολιαστεί και ότι ως εκ τούτου είναι ασφαλές το ζώο. Νομίζω ότι αυτό με μια δήλωση υπεύθυνη μπορεί να γίνει δεκτό, ελπίζω, και από τα διάφορα κράτη, μέλη. Αν και πρέπει να πω ότι δεν είμαι βέβαιος πόσο σημαντικό είναι αυτό να δείξουμε περισσότερη αυστηρότητα ή αντίθετα να περισσότερη επίοικια προς τον ιδιοκτήτη του ζώου και να πούμε ότι εντάξει έχουμε σαγαγενά κανόνα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα μελήματα που αφορούν και τον πολιτή. Άλλες τροπολογίε αφορούν τις ε, φυσικές καταστροφές. Τις έχουμε συμπεριλάβει, νομίζω το καλύπτουμε ικανοποιητικά. Υποχρέωση για ενημέρωση ενό κράτου μέλου προς την κοινή γνώμη. Για μένα είναι αυτονόητη αυτή. διάταξη δηλαδή την οποία εισάγουμε εμείς εδώ, που υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη και που λέει ότι εισάγονται κάποιοι κανόνες για τη διακίνηση των ζώων, δεν νομίζω να είναι πρόβλημα. Να λησμονήσουν δηλαδή, να ενημερώσουν τα κράτη-μέλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι περιττό, αλλά αν θεωρείτε ότι πρέπει να πει διάταξη μέσα στο κείμενο, υποχρέωση για ενημέρωση και πληροφόρηση, η οποία ή άλλω θα έπρεπε να υφίσταται, αυτονόητα δηλαδή να υφίσταται. Επίσης, πολλές είναι οι εδώ αρχίζω να είμαι και κάπως επιφυλακτικός για το αν ήταν εύστοχε. για τον ε, περιορισμό του νότα του αριθμού και τη ρύθμιση για τις παρεκκλήσεις. Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε για να αποφεύγεται και το λαθρεμπόριο και όλα αυτά, ίσχυε ότι μπορεί να μεταφερθούν μέχρι πέντε ζώντα ζώα πέραν των συνόρων. Αλλά διαρκώς ακούμε παρατηρήσεις, ε, ρωτήσεις κτλ. Ότι είναι δύσκολο να τηρηθεί αυτός ο κανόνας των πέντε ζώων και έτσι είπαμε καλώς ας βρούμε μια λύση που να επιτρέπει πιο ευέλικτες, πιο ευέλικτη προσέγγιση. Και άρα δυνατό μου φαίνεται από την πλήρη απαγόρευση μέχρι την απόλυτη ελευθερία, πάλι βλέπω τεράστιες αποκλήσεις φυσικά αποστάσεις, μπορούμε να βρούμε κάπου μια, μια λύση, στα Στα διάμεσα χρόνια θα μπορούσε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει καταθέσει και μια ε, έκθεση, πιστεύω, για το πώς λειτουργήσε το σύστημα και πόσα ζώα έχουν μεταφερθεί και όλα αυτά για να, δούμε, να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Άρα νομίζω να, θα έλεγα ότι είναι καλό να μείνει η τροπολογία μου. Άλλωστε υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες αφορούν κυνηγού και τα ζώα, τους ε, σκύλους που συνοδεύουν τους κυνηγού κτλ. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια δεν είδα από καμιά ένωση κυνηγών της Ευρώπης ή από οποιαδήποτε ένωση κυνηγών ε, μήνυμα ηλεκτρονικό ή άλλο που να μου υποδεικνύει ότι τους ενοχλούν οι ρυθμίσεις αυτές. Εν πάση περιπτώσει είναι θέματα τα οποία θέλουν συζήτηση, αλλά πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλώς για μια παρέκκληση σε περίπτωση κάποιων εκδηλώσεων που απαιτούν μεταφορά ζώων εφόσον προσφέρονται τα απαραίτητα αποδεικτικά. Τώρα, τα στοιχεία που θα μπουν μέσα στο έγγραφο ταυτότητα. Εδώ έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα προτάσεων. Νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε στο είδος του ζώου, το χρώμα, το, το τη ράτσα. Τους τελευταίους δύο κατόχους, οι ιδιοκτήτες όπως το λέγαμε, θα μπορούσαμε νομίζω να το έχουμε γιατί... Ε, αλλά δεν χρειάζεται να το γράψει μέσα στον νόμο γιατί αυτομάτως με το που γίνεται ένα ζώο ή πολίτες έναν ιδιοκτήτη και μετά αυτό μεταβιβάζεται με κάποια περαιτέρω πώληση παραμένει στα στοιχεία ταυτότητάς του πρώτος και δεύτερος ιδιοκτήτης. Για την θέση εφαρμογή τρία χρόνια μπορούμε να πούμε ναι, να αφήσουμε ένα περιθώριο τριών ετών για να μπορέσουν να προσαρμοστούν τα κράτη-μέλη και οι κτηνίατροι και όλοι αυτοί, ώστε να τηρήσουν όλε τι προτάσει. Αυτά κυρίε και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις ε, τροπολογίες που έχουν να κάνουν με άλλες διατάξεις όπως ε, θανάτωση κτλ. Καλές είναι και αυτές. Εν πάση όμως το σημαντικό είναι να έχουμε την ουσία του θέματος, να μην μιλήσουμε απαραίτητα για μια ευρύτατη βάση δεδομένων που θα καλύπτει όλα τα ζώα στην Ευρώπη. Είναι πολύ περιπλοκό, πολύ σχηδές το πρόβλημα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε μέσα σε αυτή την έκθεση και με αυτές τις τροπολογίες. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην έκθεση για την ευημερία των ζώων, όπου να, θα πρέπει να μας δώσει η Επιτροπή τις τελευταίες εξελίξεις και την αποτίμηση ως προς την υλοποίησή της και να περιοριστούμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ τώρα. Κύριο Παλάκη, Επειδή συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι περισσότερες των προτεθεισών τροπολογιών μπορούν να βελτιώσουν αυτόν τον κανονισμό. Και επομένως θα πρέπει να τις επιψηφίσουμε. Εγώ συμφωνώ με κάθε τροπολογία που θα φέρει περισσότερη διαφάνεια και που θα καταστήσει δυσκολότερο το να παρακάμπτει κανεί το σύστημα με την παραπίση και πλαστογράφηση εγγράφων και γι' αυτό σας ε, προτείνω τα διαβατήρια και τα άλλα έγγραφα που δίνουν ταυτότητα να τυπώνονται από εγκεκριμένους οργανισμούς. Εκεί θα έχουμε ε, πληροφορίες σε σχέση με τους δύο τελευταίους κατόχους του εγγράφου. Όμως θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα στα στοιχεία των προηγουμένων κατόχων σε κάποιο αρχείο. Και έτσι θα αποφύγουμε την κατάσταση κατά την οποία ε, κάποιος για πονηρούς σκοπούς θα θέλει να τα παραπείσει αυτά τα έγγραφα και έτσι θα παραποιεί τις πληροφορίες για την προέλευση του ζώου. Θα έχουμε, να έχουμε βέβαια και με ηλεκτρονική βάση δεδομένων και οι περισσότερες ε, χώρες μέλη έχουν αρκετά καλά ηλεκτρονικά συστήματα. Όμως αυτό το οποίο λείπει τώρα είναι κάποια διασύνδεση αυτών των ε, βάσεων δεδομένων ε, μέσω ενός κεντρικού συστήματος. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω την άποψη της Κομισιόν επ' αυτών. Εγώ πάντως συμφωνώ. Είμαι υπέρ της παρέκκλησης. ότι να μην ζουν για την κατοικίδια ζώα, η ζώα συντροφιάς, πώς τα λένε, ε, τεστ αντισωμάτων, σε σχέση με την είσοδο σε κράτος μέλος μέσω τρίτης χώρας, η οποία δεν έχει επαρκείς ε, κανονισμούς και ρυθμίσεις, ε, παρά μόνο ε, εάν το ζώο παραμένει σε περιορισμό σε περιορισμένο χώρο, σε κάποιο αεροδρόμιο. Όμως, να χρησιμοποιείται αυτή η, η παρέκκληση για ολικούς τρόπους μεταφοράς και έτσι κι αλλιώς τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ όσον αφορά τις οδικές μεταφορές της συνήθεις. Επομένως, σε πάρα πολύ λίγα σημεία διαφέρει είμαι από τον εισηγητή. Ας πούμε, επί πόσα χρόνια θα πρέπει να κρατούν τα στοιχεία των κατοικιδίων οι κτηνίατροι και τι να χρειάζεται ως αποδεικτικό αντικείμενο για την, ε, για την εξαίρεση σχετική με το να ταξιδεύουν πάνω από πέντε ζώα μαζί για να πάνε σε κάποια επίδειξη, σε κάποιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντέβις, εκ των Φιλελευθέρων. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ακούω ότι οι γάτες τους ήδη δεν κάθεται πάνω στο καναπέ. μου κάθεται πάνω στο πληκτρολόγιο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις απομακρύνω από εκεί. Ήθελα να αναφέρω δύο σημεία. Το πρώτο είναι το ζήτημα της κεντρικής βάσης, του κεντρικού σημείου αναφοράς. Πιστεύω στο σύνολο αυτό είναι λίγο υπερβολική νομοθεσία. Άλλοι λένε βέβαια ότι είναι εύκολη η υλοποίηση. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση της Κομισιόν σε αυτό. Αλλά προς στιγμή για μένα αυτό φαίνεται ε, μη αναγκαίο βήμα. Επίσης το ζήτημα για την εχνηλασιμότητα των ιδιοκτητών, των κατόχων, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχουμε αυτές τις πληροφορίες, να είναι. Αλλά κοιτώντα όλη αυτή την εκθέση και τις 165 τροπολογίες που υπέβαλε ο κ. Σνέλχαρντ, αυτό που με ανησυχεί κυρίω είναι θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο κανονισμός θα είναι εύκολος στην υλοποίηση, στην εφαρμογή, και ότι θα παρέχει αποτελεσματικέ διασφαλίσεις κατά τη λύσας. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι δεν αφήνουμε κενά παραθυράκια για την εμπορική μετακίνηση των ζώων και απαράδεκτες πρακτικέ. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια μερίδα εδώ στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τη μεταφορά εξωτικών ε, ζώων συντροφιά. Καταπληκτική ημερίδα. Αυτά τα ζώα συχνά συλλαμβάνονται στην αγρεφήση σε περιοχέ γύρω από τον Ισημερινό συνήθω όπου υπάρχει τεράστια βιοποικιλότητα. Δεν υπάρχει βέβαια απειλή εκεί για τη Λύσα, αλλά τα νούμερα που είδαμε και οι φωτογραφίε 70% των ζώων πεθαίνουν ήδη ε, στη φάση του χονδρικού εμπορίου, πριν φτάσουν καν στα καταστήματα. Αναρωτιόμουν λοιπόν κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να ε, αναφέρουμε και αυτό το ζήτημα μέσω κάποιες τροπολογίες, γιατί αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε εδώ, αυτό που είναι σημαντικό, βασικά σκεφτόμαστε για σκύλους, γάτες, ε, και δεν θέλουμε να έχουμε και προβολικό κρατικό έλεγχο, διότι ο κόσμο αγαπάει τα ζώα συντροφιά και αυτοί που τα πουλούν τα αγαπάνε, αλλά καθίστε σαφέ από την παρουσίαση ότι όταν είναι να βγάλει κάποιο χρήματα, δεν δίνει δεκάρα για τα ζώα δεν είναι παρά κομμάτια κρέας από τα οποία βγάζει κάποιος ε, χρήματα. Ήθελα λοιπόν να, να μας πει η Κομισιόν, καταλαβαίνω ότι αυτό το ζήτημα είναι ε, επιπρόσθετο, δεν είναι... Ε, υπάρχει κάποιο σχέδιο της Κομισιόν για τα εξωτικά ζώα και για το εμπορίο τους στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ Chris Davis, ε, Jill Evans για τους πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι μεγάλη πρόκληση το να επιτρέπουμε τον κόσμο να κυκλοφορεί με τα ζώα συντροφιά του, αλλά ταυτόχρονα να ε, φροντίζουμε και για την ε, δημόσια ασφάλεια και για τα ζητήματα δημόσιας υγείας. Πιστεύω ότι έχει προσδιορίσει τα κυριότερα ζητήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να επικεντρωθούμε επειδή όλοι έχουμε ως κοινό στόχο να επιτύχουμε αυτή τη σωστή ισορροπία και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη βάση δεδομένων, φοβάμαι πως δεν μπόρεσα να παραστώ στη ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, αλλά φυσικά αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες που αφορούν την γραφειοκρατία και συμφωνώ με αυτές τις ανησυχίες σε κάποιο βαθμό, αλλά από όσο κατάλαβα, Υπάρχει ήδη κάποια μορφή εθνικής βάσης δεδομένων σε 26 κράτη-μέλη. Συνεπώς, ε, έχει νόημα να συντονίσουμε αυτές τις βάσεις δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερη ειχνηλασιμότητα, ταχύτερη αντίδραση σε οποιαδήποτε κρούσμα νόσου. Θα μπορέσει επίσης να βοηθήσει να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για να καταφέρουμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε από τον εισηγητή είναι η εμφύτευση των πομποδεκτών. Το μόνο πρόβλημα που φαίνεται να απομένει εδώ είναι κατά πόσο θα πρέπει να επιβλέπεται αυτή η ενέργεια από κάποιον κτηνίατρο. Αυτό που με ανισχύει εμένα ε, γνωρίζω εγώ ότι στην Ουαλία οι οργανισμοί ευημερίας των ζώων και οι τοπικές αρχές ε, πραγματοποιούν αυτή την ενέργεια σε παντός είδους χώρους και υπάρχει πάντα και η απέτηση του να υπάρχει πάντοτε κτηνίατρος μπορεί να παρεμποδίσει αυτή τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους και οδησυγητές το ζήτημα του μέγιστο αριθμού πέντε ζώων. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του Κρίς ότι θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση αυτού του μέτρου, αλλά από την άλλη όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα εδώ. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Παρομοίως ε, και με την παρέκκληση για τα ζώα ηλικία κάτω των τριών μηνών. Ε, αυτό που είναι σχεμένα είναι ότι είναι αυτά που ανέφερα και την τελευταία φορά που συζητήσαμε αυτόν τον κανονισμό ε, Αναμένω λοιπόν να συζητήσουμε αυτέ τι ιδέε μεταξύ σχεδόν εισηγητών και είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε συμφωνία στα περισσότερα, ενώ σε όλα από αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφο Κουλέκη. Αλλά θα, τα, θα την εκπροσωπήσει κυρία Ρόσπαχ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω ένα έγγραφο της κυρίας Γιανακουδάκη, σκιώδους ηγετρίας για το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα σας το παρουσιάσω στα αγγλικά. First of all... Πρώτα πρώτα θα πρέπει να δεχθούμε ότι βελτιώνει σωστές προτάσεις του της πρώτης Κομισιόν και αυτό θα πρέπει να δούμε είναι το πώς θα ισχύσουν αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής όσον αφορά τα μικρά κτηνιατρία και θα πρέπει να περιορίσουμε αυτή τη δεκαετία των, των μικροτσίπ στους κτηνίατρους και θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές, τα ελάχιστα πρότυπα και για τους υπόλοιπους οι οποίοι συμβάλλουν σε τη διαδικασία. Επίσης, αυτό που θέλουμε είναι το να καλύψουμε το ότι πρέπει να συνεχιστεί η ελεύθερη διακίνηση των κατοικιδίων σε αυτές τις διάφορες εκδηλώσεις όπως ε, αυτοί οι διαγωνισμοί σκύλων. Να μην παραβλάψουμε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει όμως να εμποδίσουμε και τις ε, απάτες σε σχέση με το άρθρο 40 και να καταστεί ξεκάθαρο ότι στην περίπτωση των κατοικιδίων που έχουν περάσει από τους σχετικούς ελέγχους την ευθύνη την έχει ο Κύριος να το επιστρέψει στη χώρα προέλευσης το ζώο, όπως ακριβώς λέει και η τροπολογία μας το άρθρο 37. Παρ' αυτά, συνολικά, θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης και οι πρώτες κομισιόν είναι αξιόλογες και να δούμε πώς σε συνεργασία με τον εισηγητή θα μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιους συμβασμούς στην Επιτροπή πριν την Ολομέλεια. Αυτά από πλευρά μα. Αλλιώ, όπω και ο Κρίτς, και ο έχω και εγώ και σκύλο και γάτα που ξαπλώνουν όπου τους γουστάρει. Και δεν θα φανταζόμουν ποτέ να τους περιορίσω. Μου φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το υλοποιήσουν αυτό οι κτηνίατροι καταρχά εν γέννη. Και τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εγώ. Μεγάλη σημασία έχει να εκπαιδευτεί ο κάτοχος ενός ζώου, να έχει την ευθύνη του στην πραγματικότητα. Γιατί αν κανείς δεν είναι υπεύθυνο, εάν δεν φροντίζει να πάει να εμβολιάσει, να βάλει το ενότιο ή τον ε, ε, αναμεταδότη στο ζώο, δεν χρειάζεται να έχει ζώο στο σπίτι του, εάν δεν μπορεί να συμπεριφέρεται υπεύθυνα. Νομίζω ότι όσο δύσκολε και είναι οι συνθήκε καμιά φορά, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε ένα ζώο έχουμε και τι σχετικέ ευθύνε. Ευχαριστώ. Η Γιούτα δεν είναι εδώ. Κύριε Σανώνη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή για τη δουλειά του. Είναι ένας κανονισμός πολύ σημαντικό όλο αυτός, διότι προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να μεταφέρουν τα ε, δικά του ζώα εντός τη ευρωπαϊκή Ένωση Αφορά επίσης και την προστασία της ευημερία των ζώων, αλλά και την προστασία της υγεία των πολιτών κατά αυτών των ε, εύκολα μεταδεδομένων νόσων όπως η Λύσα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων, που ενδεχομένως θα είναι προσπελάσιμη εύκολα από όλα τα κράτη-μέλη, ο εισηγητής παρατήρησε ότι ε, είναι γραφειοκρατία. Φυσικά αυτό το σύστημα του microchip, ε, ε, αυτά τα συστήματα microchip και βάση δεδομένων υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη σε πολλές ε, περιοχές της Ιταλίας έχει οθετηθεί αυτό το σύστημα. Ε, διαβεβαιώ τον συναδέλφο ε, ότι αν κάποια ηλικιωμένη κυρία πρέπει να μεταφέρει τη γάτα της σε ένα άλλο κρατός μέλος θα έρθει σε επαφή με κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο όπως θα κλείσει το ξενοδοχείο μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου και το εισιτήριο μπορεί να παρέχει να προμηθευτεί τα ίδια γραφά και για το ζώο της φυσικά. Αυτό που με ανισχύει εμένα προσωπικά είναι ότι προβλέπονται αυτές οι παρεκκλήσεις όσον αφορά τους εμβολιασμού για τη Λύσα και ο συνάδελφος ε, δικαίως υπενθύμησε ότι υπάρχουν παραθυράκια μεταξύ των 12 και 16 εβδομάδων όπου τα κουτάβια είναι ανοσοποιημένα χάρη στη μητέρα αλλά πρέπει να φροντίσουμε να διαβεβαιώσουμε το εξή. Υπάρχουν ελάχιστοι έλεγχοι στα σύνορα σχεδόν ποτέ δεν ελέγχονται τα ζώα που μεταφέρονται. Εάν πρόκειται λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν κανονισμό πιο ελεύθερο από αυτό που υπάρχει, πρέπει να πούμε ότι στην Ιταλία υπάρχουν ε, διοικητικές και ποινικέ κυρώσεις ε, για τη μεταφορά ε, ζώων, ας πούμε κουταβιών μικρότερων, νεαρότερων των τριών μηνών. Επίσης υπάρχει το θέμα του παρανομεμπορίου που ανθεί Μόνο στους τελευταίους 5-6 μήνες ε, στην Ιταλία κατασχέθηκαν στα βορειοανατολικά πάνω από 400 κουτάβια ξεχωριστά από την Ουγγαρία, από εκτροφή στην Ουγγαρία και το ε, περισσότερα είχαν παραποιημένα έγγραφα και τα περισσότερα ήταν πολύ μικρότερα από τριών μηνών. Το πρόβλημα λοιπόν των λοιπόν ελέγχων θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να ε, έχουμε μία, πιο αυστηρούς κανόνες και όχι, πιο, και όχι λιγότερο αυστηρούς. Όσον αφορά την τροπολογία 34 του συντάκτη, οι παρεκκλήσεις για ε, πάνω από πέντε ζώα, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε, διότι και αυτό αφήνει περισσότερες ελευθερίες σε όσους θέλουν να καταχραστούν αυτή την νομοθεσία. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη σκέψη που αφορά Ορισμένες τροπολογίες αναφέρομαι στην 181, 190 και 219. Εδώ μιλάμε για συνοδευτικά έγγραφα για ζώα του μέρους Β του παραρτήματος 1 που δεν είναι ούτε γάτες, ούτε νηφίτσες, ούτε σκυλιά. Ειδικότερα ε, πτηνά. Και εδώ προτείνονται τροπολογίες που για μένα είναι ανησυχητικέ. Διότι πρώτα απ' όλα θέλουν να καταργηθεί ο περιορισμός των πέντε ζώων και να μην υπάρχει ε, όριο σε αυτή την περίπτωση. Επίσης ε, μιλάνε επιπλέον για συλλογικές άδειες, όχι επιμέρους άδειες. Δηλαδή ίσως δεκάδες πτηνά που μπορούν να μεταφερθούν με ένα μόνο έγγραφο. Ενδεχομένω πολλών ιδιοκτητών προσοχή λοιπόν σε αυτό, διότι ε, Μία από τι αιτίε για την οποία υποβάλλονται, υποβάλλονται τέτοιε τροπολογίε είναι για να υποβάλλονται σε ελέγχου υγειονομικού τα πτηνά. Άλλη μία περίπτωση που είχαμε στην Ιταλία, είχαμε μια επιδημία της των, ε, επιδημία των πτηνών. Αποφασίστηκε να θανατωθούν πάνω από 40.000 ε, πτηνά ε, εκτροφείου αλλά και καλοπιστικά και τα, οι κανόνες που προβλέπονται από τροπολογίες σαν αυτές ε, δεν πρέπει να περάσουν διότι αντικείνται στα συμφέροντα των ε, πολιτών οι οποίοι και αυτοί πρέπει να προστατεύονται από υγειονομική άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνουμε για να τους ε, για να ακούσουμε τους συναδέλφους από τις ομάδες. Εάν θέλετε, παρακαλώ, η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να παρατηρήσω ένα πράγμα. Την ιστορία λίγο αυτού του κανονισμού. Αυτός ο κανονισμός ε, αποσκοπεί στο να προλαμβάνει τη διάδοση ε, ασθενειών των ζώων, σοβαρών ασθενειών, σοβαρών νόσων, που έχουν επιπτώσεις και για την ανθρώπινη υγεία μέσω της ε, μη εμπορικής μεταφοράς ε, ζώων συντροφιάς. Αυτό το επιχείρημα ήταν δύσκολο στη μελέτη πριν από 10 χρόνια όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υιοθέτησαν τον τρέχοντα κοινωνισμό. Χαίρομαι που ακούω ότι σήμερα κατά τη συζήτηση το θέμα της διάδοσης των νόσων των ζώων μέσω της μετακίνησης ζώων συντροφιάς ε, αντιμετωπίστηκε μόνο κατελάχιστον. Γιατί, διότι ο κανονισμός πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχαν τεθεί. Δηλαδή την πρόληψη της διάδοσης των νόσων των ζώων, ε, μέσω των ζών συντροφιάς και της απλούστευσης της μετακίνησης αυτών των ζώων συντροφιάς από τους εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδεύουν με το σκυλί ή με το η γάτα τους. Έτσι λοιπόν ήθελα να παρατηρήσω ότι ο τρέχον κανονισμός λειτουργεί μια χαρά. Κατάφερε να επιτύχει τους κυριότερους στόχους του. Σήμερα ακούσαμε διάφορες παρατηρήσεις από τα μέλη του Κοινοβουλίου που ακούσαμε, αλλά που ουσιαστικά αφορούν λεπτομέρειες. Και αυτό φυσικά μας χαροποιεί το να ακούμε όλα αυτά τα σχόλια, όλες αυτές τις απόψεις και βλέπουμε ευνοϊκά την ψηφοφορία από την παρούσα και στη συνέχεια από την Ολομέλεια. Ωστόσο, όπως και να έχει μιλάμε για λεπτομέρειες ε, σε σύγκριση με το πραγματικό πρόβλημα. Και σίγουρα επαναλαμβάνω ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα απλά, να μην τα περιπλέκουμε. Εκτός εάν έχουμε εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο, οφείλεται, το οποίο προκύπτει από τους ε, σημερινούς κανόνες. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα, όπω γνωρίζουμε, είναι το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν παράνομες μετακινήσεις ζώων που διατίθενται στο εμπόριο αλλά που στην ουσία μεταφέρονται με βάση κανόνες ε, μη εμπορικούς για μεταφορά ζώων. Και εκεί το θέμα είναι το θέμα ελέγχων. Ε, ελέγχοι που είναι αρμοδιότητα των κρατών μέλων και που μέσω του άρθρου 35 έχουμε ενισχύσει στο άρθρο 35 δηλαδή της πρότασης της Κομισιόν ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη ώστε να διεξάγουν αυτούς τους ελέγχους. Συζητήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τη χρησιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τελειοποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μη εμπορικών μετακινήσεων ζώων συντροφιάς ε, μεταξύ κρατών μελών. Δηλαδή το αντικείμενο του σκοπός τους είναι διαφορετικός από το σκοπό του παρόντος κανονισμού. Το να εναρμονίσουμε λοιπόν στο εσωτερικό του παρόντος κανονισμού αυτού του είδους της βάσης δεδομένων μου φαίνεται για αυτό το λόγο ακατάλληλο. Θεωρώ ότι θα οδηγούσε σε περιττή γραφειοκρατία και δεν θα προσέχετε απόψη ασφάλεια ε, των μετακινήσεων. Δεν θα προσθεθεί τίποτα από άποψη ασφάλεια των μη εμπορικών μετακινήσεων. Αναφέρθηκε ένα πρόβλημα σε σχέση με τα ζώα συντροφιά, τα εξωτικά ζώα συντροφιά. Και εδώ ρωτήθηκε η Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με τις εισαγωγές. Και σε αυτή την περίπτωση οι εισαγωγές είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν εμπίπτει ε, στο νομικό πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αλλά έχουμε προτάσει στην Κομισιόν ε, τις οποίες συζητάμε στο πλαίσιο της ε, μόνιμης επιτροπής και κυρίως για κάποια ζώα που θέτουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το συχνότερο όμως πρόβλημα είναι Ποιο είναι ο σκοπό, ο απότερο σκοπό είναι η ευημερία των ζώων ή η υγεία των ζώων, διότι δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά του τελικού σκοπού Προσπαθούμε να προλαμβάνουμε ασθένειε ή προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι τα ζώα θα ταξιδεύουν με υποσυνθήκες τέτοιες ώστε να μην υποβαθμίζεται η ευημερία τους. Πάντα θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτών των διεπιχειρημάτων. Διαφορετικά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεχώς προβλήματα νομικής βάσης, αναλογικότητας κτλ. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό. Όσον αφορά η Κομισιόν διατηρεί αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό το τρέχον νομικό πλαίσιο. Υπενθυμίζω ότι η κύρια αιτία της πρότασης αυτής ε, από την Κομισιόν ήταν η ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή να μην γίνουν σημαντικέ τροπο, ουσιώδεις τροπολογίες στο τρέχον νομικό πλαίσιο. Επ' αυτού σας υπενθυμίζω τους υπάρχοντες κανόνες σε σχέση με τη μετακίνηση άνω των πέντε σκυλιών, γατών και ε, νηφίτσων, νηφιτσών. Όταν ένας ιδιοκτήτης θέλει να μετακινήσει, χρειάζεται να μετακινήσει Α, πάνω των πέντε τέτοιων ζώων οι κανόνες που έχουν εφαρμογή είναι οι κανόνες των εμπορικών ζώων της εμπορικής μετακίνησης ζώων δηλαδή τα εν λόγω ζώα ναι, ναι. πρέπει να πιστοποιηθούν από κτηνίατρο το ε, πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια και εφόσον ισχύει το πιστοποιητικό μπορούν να μετακινηθούν τα ζώα αυτά από το ένα κράτος στο άλλο χωρίς μεγάλες δυσκολίες αλλά χρειάζεται κτηνιατρική πιστοποίηση, χρειάζεται αναγνώριση, ταυτοποίηση των ζώων και όλα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω κανονισμού της Κομισιόν. Το κανονισμό 388 του 2010. Η Κομισιόν ζητάει από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τις εγχωρήσουν κατά το δικαίωμα κατά εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 40, παράγραφος 2, όπου η Κομισιόν βάσει εμπειριών που έχουν ήδη εμφανιστεί μετά από τα δύο χρόνια υλοποίησης του κανονισμού που αναφέρθηκε θα θεωρήσει σκόπιμο να επικυρώσει τους υπαρχόντες κανόνες. Αλλά εδώ μιλάμε για λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι εμείς ως Κομισιόν θα επικυρώνουμε το αίτημα προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μας εκχωρήσουν ε, τη δυνατότητα κατεξουδότησης πράξεων για τη ρύθμιση του θέματος αυτού. Όσον αφορά την εμφύτευση των transponder, τα microchip. Και εδώ επικυρώνουμε τους τρέχοντες κανόνες που φαίνεται να λειτουργούν. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε άλλη γραφειοκράτεια. Αφήνουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ποια είναι η ιδανική, ο ιδανικός, ποιος είναι ο ιδανικός φορέας ε, για να διενεργεί αυτή την επέμβαση. Πιστεύω ότι αναφέρθηκα στα κυριότερα σημεία, αλλά και άλλο ένα, ο κανονισμός. Δεν έχει τη φιλοδοξία να εχνηλατεί τέλεια κάθε σκύλιο και κάθε γάτα που μετακινείται από ένα κράτος σε ένα άλλο. Το να, επιτευχθεί τέτοια χνηλασιμότητα, η επίτευξη τέτοια χνηλασιμότητας χρειάζεται τεράστιο κόστος και τεράστιο έργο δυσανάλογο σε σχέση με τους στόχους του κανονισμού. Υπενθυμίζουμε ότι σε τεράστιο βαθμό ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί με τους τρέχοντες κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα παρακαλώ τον κύριο Σνέλχαρτ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι για τα σχόλια στην έκθεση και πιστεύω ήταν πολύ χρήσιμες και οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συζήτηση. Θέλω απλώ να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να λησμονούμε για ποιο λόγο, ποιον λόγο εισάγεται αυτή η νομοθεσία και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα που θέλουμε. Και να αφήσουμε αυτά τα οποία δεν έχουν θέση να επιληθούν εδώ προκύπτει και από τις συνομιλίες με τους κοιόδης ηγητές. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε μια ευρύτατη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σνέλχαρτ. Έξι Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία των δύο αυτών εκθέσεων. Ε, προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών δεν έχουμε ορίσει. Κλείνει το θέμα αυτό προς το παρόν. Και έτσι περνάμε στο 21. Και παρακαλώ την ομάδα των Πρασίνων να λάβει το λόγο η κυρία Χάση. Α, όχι, πρώτα η Επιτροπή παρακαλώ. και ευχαριστώ πολύ που σπεύσατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πλήρως τους κινδύνους αυτών των υγειονομικών προβλημάτων, των προβλημάτων υγείας που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση του πετρελαίου ντίζελ και αυτά τα ξέραμε πριν καν προκύψει αυτή η έκθεση της 12 η Ιουνίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας γιατί ήδη Είχαμε δηλαδή κάποια πρωτοβουλία πριν κάνει εγκριθεί αυτή η εκθέση, ώστε να μειώσουμε τι επιπτώσει από τι ε, εκπομπέ των, των για, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο diesel. Και πρόκειται για την νόρμα Euro 6 που θα αφορούσε τα, τα φορτηγά ε, Euro 5, Euro 6 και με αυτόν τον τρόπο είπαμε ότι στο εγγύς μέλλον πρόκειται να έχουμε μείωση πολύ των ε, εκπομπών αυτών των οχημάτων. Η αποστολή μας είναι εξή. Θέλουμε να έχουμε σημαντικές μειώσεις στο μέλλον από το 2014 για τα αυτογίνητα και έτσι να μειώσουμε σημαντικά τις επιπτώσεις της υγείας των εκπομπών αυτών. Για φορτηγά και, και νταλίκες. Έχουμε τώρα την, ε, την εφαρμογή και την τοποθέτηση καινούριων ε, ανταλλακτικών και εξαθμίσουν σε αυτά, ούτω ώστε να οδηγηθούμε σε κάποιο είδου ε, ε, μείωση των εκπομπών και το 2013 ήδη να, να ολοκληρωθεί όσον αφορά τα φορτηγά και να προχωρήσουμε μετά στις συνταλίκες. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε σε, μείωση αυτών των εκπομπών και και αυτόν τον τρόπο να έχουμε τη μείωση αυτών των μορίων των σωματιδίων. Με λίγα λόγια, έτσι θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές αυτών των σωματιδίων από τους κινητήρες πετρελαίου ντίζελ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της. κυρία Χάση, αλλά εάν κατάλαβα καλά, εσείς αναφερθήκατε μόνο στις προδιαγραφές εκείνες που ήδη έχουν ε, εγκριθεί. Πρόκειται τώρα για νέο κατάταξη των ε, αερίων εκπομπής εξάτμισης τέλος πάντων αυτών των οχημάτων που και θεωρήθηκαν καρκινογόνα όμως γνωρίζετε ότι θα πρέπει να δούμε διάφορα στοιχεία, τη εθνισμότητα, το κόστος της, ε, του καθαρισμού των εκπομπών και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως πρόγραμμα το να κάνει κάποια επικαιροποίηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους. για αυτές τις εκπομπές. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον υπάρχει το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του να αλλάξει αυτά τα πρότυπα εκπομπών των οχημάτων. Τέλος πάντων αναφέρουμε σε αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί. Αλλά θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε ασφαλέστερα τα πρότυπα τα οποία ήδη έχουν έχει αποφασιστεί. Ευχαριστώ. Κορίν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η σάτουχάση συνάδελφος, γιατί αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Οπότε το να κάνουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές είναι σημαντικό. Αλλά η εφαρμογή των ισιών των κανόνων και καθώς και κάποιες κυρώσεις που πρέπει να προβλέπονται και το οποίο αυτό το είναι καυτό ζήτημα για τη χώρα από την οποία προέρχομαι. Δεν τηρούνται οι υπάρχοντες κανόνες και άρα και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι κοστίζει πάρα πολύ στο κράτος ε, το τι γίνεται, αυτές οι ασθένειες οι αναπνευστικές από αυτά τα λεπτά μικρά σωματίδια Άρα θα πρέπει να αναλυφθεί δράση κατεπίγουσα για το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Έχουμε στην επικαιρότητα της επόμενης χρονιάς το θέμα των, ε, του καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν νέες προτάσεις για τις οριακές τιμές. Στο παρελθόν ορίζαμε στόχους Νομίζω ότι μπορούμε πια να είμαστε και πιο φιλόδοξοι. Διαπιστώνουμε όμως ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των πηγών, ορίζοντας οριακές τιμές. Δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα των, της πηγής της ρήπανσης και νομίζω καλό θα ήταν να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. επιδιώκοντας χαμηλότερη κατανάλωση, η οποία μοιραία οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές. Αλλά βέβαια αυτό απαιτεί πιο πολλά χρήματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια λογική ανάλυση κόστους και αποτελέσματος. Χρειάζεται να επιμείνουμε πολύ σε αυτό. Καλή λοιπόν η πρόταση. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Αλλά ο κύριος Σλίτερ έχει στο λόγο, παρακαλώ. Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι όταν ήμουν στη χώρα μου και συνάντησα ειδικού για το περιβάλλον, όλοι συζητούσαν για τα πρότυπα σωματιδίων στον αέρα και αναρωτιούνται δεν θα προταθεί καμία, κανένα πιο αυστηρό όριο, διότι αυτό είναι ανησυχητικό. Ε, είναι πιο καρκινογενή αυτά. Ποια είναι η θέση σας για το PM1 και τα μικρότερα σωματίδια. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στείλει άλλο το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή να ξαναπάρει το λόγο. Για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πολλά υπόθηκαν. Όσον αφορά τη στρατηγική για την ποιότητα του αέρα, όπω κατάλαβα εγώ, ο κ. Ποτότσνικ, επίτροπο για το περιβάλλον, προτίθεται να προτείνει το 2003 αναθεώρηση τη στρατηγική ποιότητα του αέρα. Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, δηλαδή τα αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση τη ε, στάθμη των ε, ε, ρηπογόνων σωματιδίων έχουν ληφθεί πρωτοβουλίε, είναι αλήθεια, ορισμένα Μέτρα λήφθηκαν πρόσφατα και στον τομέα των, της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τομέα των φορτηγών. Ε, εισάγονται προοδευτικά, ειδικότερα για τα αυτοκίνητα, διότι από το 2014 θα τεθεί σε ισχύ ο κανόνας που θα υποχρεώνει τη χρήση φιλτρού σωματιδίων. Αυτό το φίλτρο σωματιδίων το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη και το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω της σημαντικής μείωσης τόσο της μάζας της ποσότητας δηλαδή των σωματιδίων. Έχουν ήδη προβλεφθεί προδιαγραφές αλλά και μέτρα, αλλά αυτά θα τεθούν ε, σταδιακά σε ισχύ. Στη διάρκεια των συζητήσεων για τις διάφορες αυτές πρωτοβουλίες, ε, εδώ μάλιστα σε αυτή την αίθουσα συζητήθηκε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους τρέχοντες στόλους, διότι ξεκινάμε από την αρχή ότι ένας στόλος αυτοκινήτων ή φορτηγών ανανεώνεται κάθε 8 χρόνια και συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του retrofitting, της αναβάθμισης του υπάρχοντος στόλου, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες ειδικότερα φορτηγών που χρησιμοποιούν δίζελ, να τα εξοπλίσουν, τα φορτηγά αυτά, με εξοπλισμούς που θα μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές και ειδικότερα σωματιδίων. Και αυτό το μέσο βρίσκεται υπό προετοιμασία. Το τελευταίο μέσο που βρίσκεται υπό προετοιμασία είναι η μείωση ε, των σωματιδίων από τα εργοταξιακά μηχανήματα. Εδώ μιλάμε για νέες ε, προτάσεις ε, που σημαίνει ότι το 2013 θα συμπληρώσει τη μείωση των σωματιδίων στην πηγή από τους διαφορούς τομείς δραστηριότητας. Τώρα η ερώτηση το κατά πόσο θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τις μελέτες αντικτύπου ή ωφελών που έγιναν για τις ε, σημερινές προτάσεις ε, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα νέα στοιχεία είναι μια δυνατότητα. Δεν είναι κάτι που έχουμε ενσωματώσει ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση τις νέες μελέτες αντικτύπου, ειδικότερα αυτές για τα εργοταξιακά μηχανήματα, τα non-road mobile machinery, δηλαδή το σύνολο χρησιμοποιούνται για τα μηχανήματα που δεν κινούνται σε δημόσιες οδούς. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και ε, όταν θα ολοκληρωθεί σε λίγο η μελέτη αντικτύπου. Αυτά τα στοιχεία μπορούσα να σας παρέχω για να διευκρινίσουμε λίγο ή να διασαφηνίσουμε λίγα τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τη ευκρίνηση. Έχουμε βέβαια σημαντικές πρόοδους όσον αφορά την ε, μάζα των ε, μικροσωματιδίων. Τα μικρότερα έχουν ιδιαίτερη σημασία, αυτά τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν στους, στις κυψέλιδες του πνεύμονα. Ασφαλώς με ρημνά για καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και εμείς. Ευχαριστώ πολύ για την ευελιξία σας. Βλέπω να έχουμε ολοκληρώσει το θέμα αυτό και πάμε στο σημείο υπαριθμών 20. Μια ανταλλαγή απόψεων από τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Χάντζεν που με ιδιαίτερη ευελιξία ήρθε στην Επιτροπή να μας μιλήσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου επιτρέπετε να κάνω μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις ε, για την πρόσφατη ανακοίνωσή μας. Χάρηκα ιδιαίτερα που δείξατε ευελιξία και μπορέσατε να μου αφιερώσετε κάποιο χρόνο σήμερα αντί για αύριο. Ευχαριστώ. Εμείς ε, δημοσιοποιήσαμε μία ανακοίνωση για την τοξικότητα των χημικών μειγμάτων και ειδικότερα για τις ε, επιδράσεις των συνδυασμών χημικών και αυτό που θα κάνω θα είναι να σας συνοψίσω τους δύο πυλώνες ε, πάνω στους οποίους οικοδομήσαμε αυτή την ανακοίνωση. Και μετά θα σας δώσω μία παρουσίαση των γενικότερων δράσεων που θεωρούμε απαραίτητο να παρακολουθούμε. Αρχικά διενεργήσαμε μία μελέτη υψηλού επίπεδου για την τοξικότητα των μεγμάτων. Αυτή την έκθεση την υποβάλαμε σε αναθεώρηση από τις επιστημονικές μας επιτροπές στη Γενική Διεύθυνσή μας για την Υγεία και βάσει του αποτελέσματος αυτής της αναθεώρησης της αρχικής μας έκθεσης προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τις επιστημονικές αποδείξεις, τα σημεία όπου υπάρχουν κενά και τα σημεία όπου θα μπορούσαμε να αναλάβουμε δράση για να καλύψουμε τα κενά αυτά. Στα συμπεράσματα λοιπόν της ανακοίνωσης ε, ε, αναφέρουμε την ανάγκη πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά γνώσεων που έχουμε, δηλαδή ειδικότερα θέλουμε να ε, αναπτύξουμε μια πλατφόρμα για, ε, με στοιχεία χημικής παρακολούθησης, ένα μέρος δηλαδή ενιαίο όπου μπορούμε να ανακτάμε πληροφορίες για τα χημικά που, παρακολουθούνται στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους και στα διάφορα ζωικά και φυτικά είδη. Αυτό θα μας δώσει κάποια εικόνα των χημικών που πράγματι υπάρχουν στο περιβάλλον και ειδικότερα των συνδυασμών χημικών που παρατηρούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας δεύτερης δράσης επιθυμούμε να εξετάσουμε το πώς θα κατανοήσουμε την τοξικότητα των χημικών καλύτερα, ειδικότερα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Έτσι, ώστε να δημιουργήσουμε μια γνωσιακή βάση η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα χημικών για τα οποία δεν συλλέγει επαρκή δεδομένα η τρέχουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια έχουμε προβλέψει δύο δράσεις που σχετίζονται περισσότερο με την νομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρώσουμε μετά από αυτές. Η πρώτη δράση αφορά ουσιαστικά το να καθίσουμε κάτω και να εξετάσουμε τα ε, χημικά μείγματα που, στα οποία έχουμε δώσει προτεραιότητα γιατί έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για αυτά και να εξετάσουμε κατά πόσο πράγματι υπάρχει ε, κίνδυνος από το εκάστοτε μείγμα και να δούμε ποια είναι τα καλύτερα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε και στο πλαίσιο ποια νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε τον αναγνωρισμένο κίνδυνο. Μια άλλη δράση που θα αναλάβουμε θα είναι να αναπτύξουμε καθοδήγηση στο πλαίσιο της υπάρξης νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των διαφορών μειγμάτων και έτσι να υιοθετήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση για την αξιολόγηση των μειγμάτων. Αυτές οι δύο τελευταίες δράσεις ε, θα καθοδηγηθούν από μια ομάδα, έτσι έχουμε αποφασίσει, από ειδικού από τις διάφορε γενικέ διευθύνσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τα χημικά, καθώ επίσης και από τους διαφόρους οργανισμούς και αρχές ε, που έχουν κάποιο ενδιαφέρον ειδικότερα για την αξιολόγηση των χημικών και ειδικότερα των μειγμάτων και των συστατικών τους. Αυτό πιστεύω σας δίνει μια σύντομη παρουσίαση της ε, ανακοινωσή μας. Ε, είμαι διατεθειμένος να ανταλλάξουμε απόψεις και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω τις, ε, ικανοποιητικά τις ερωτήσεις που θα έχουν τα αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία έχεις το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μελέτησα πολύ στενά αυτό το ζήτημα. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το μόνο που μας ανησυχεί, που ανησυχεί εμένα, είναι η ταχύτητα. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Γνωρίζουμε ότι καθυστερεί τα υπόλοιπα μέτρα. Έχουμε μια αρχή πρόληψη στην νομοθεσία μας, δηλαδή ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα ακόμη και αν δεν έχουμε 100% των απαραίτητων γνώσεων, εφόσον πιστεύουμε ότι υπάρχει απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Για αυτό το λόγο θα ήθελα να κάνω μία πρόταση για το Συμβουλίο Υπουργών των Βορείων Χωρών όπου λέει ότι επειδή τα χημικά καλύπτονται από διαφορετικές νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Υπουργών των Βορείων Χωρών προτείνει οι τιμές κατοφλίου να μειωθούν διότι η συνολική ποσότητα χημικών ρυθμίζεται σε πολλά διαφορετικά έγγραφα, ώστε να μειωθεί η έκθεση, για να μειωθεί η έκθεση σε αυτά τα χημικά πρέπει να μειώσουμε τα κατοφλία στο 10% για παράδειγμα του, της αποδεκτής τιμής ε, στις υπάρξεις νομοθεσίες ώστε το σύνολο, η συνολική έκθεση να είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη σημερινή. Αυτό θα ήταν ένα τρόπο ε, αποτελεσματικό και ω προ το κόστο για να επιλύσουμε το ζήτημα. Δεν χρειαζόμαστε νέε μελέτε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αντιμετωπίσουμε πολύ ικανοποιητικά το ζήτημα αυτό με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι με μία κίνηση να επιτύχουμε πολύ υψηλότερο επίπεδο ασφάλεια. Αναρωτιέμαι κατά πόσο η Κομισιόν ε, έχει υπόψη τη μια τέτοια λύση. Έχω και δύο ερωτήσει, ίσω λίγο χαζέ ή λίγο απλοϊκέ. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, την ισχύουσα νομοθεσία, τις διάφορες επιμέρους νομοθεσίες, μπορείτε να λάβετε υπόψη τις επιδράσεις των συνδυασμένων χημικών. Υπάρχει τρόπος να μπορείτε να ε, τις διαπιστώσετε και να ορίσετε τιμές οριακές. Εφόσον αυτό είναι δυνατό, υπάρχουν παραδείγματα όπου έχουν γίνει τέτοιες εκτιμήσεις, όπου διάφοροι έχουν λάβει υπόψη μελέτες που δείχνουν συνδυασμένες επιδράσεις χημικών και όπου έχει προταθεί η σταδιακή εξάλληψη κάποια ουσία ή έχει οριστεί κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο έκθεση. αυτη είναι η ερωτηση μου. Ευχαριστώ. Euh, ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει αναλάβει αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό συμβαδίζει με τη βούληση πολλών από εμά να συνεργαστούμε με τη Γενική Διεύθυνση για να επιτύχουμε το περισσότερο δυνατό, το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα, βάσει της, ε, των συμπερασμάτων τη ανακοίνωσή σα του Μαΐου 2012, έχω μια σειρά ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα, λέτε ότι θα υπάρχει μια αντόκομα εργασία με εκπροσώπου των αρμόδιων αρχών και των ε, οργανισμών. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι διασφαλίζει την ε, εγκάρσιο χαρακτήρα. Θα, θα, θα συνεργαστούν επίσης και οι ενδιαφερόμενοι, μη κάπα οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και θεωρείται ότι αυτή η αντόκομα δεργασία θα μπορεί να ε, αναφέρει τακτικά στο Κοινοβούλιο για την εξέλιξη των εργασιών της. Δεύτερον, η Κομισιόν προβλέπει την ε, εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για να προωθήσει μια συνεκτική αξιολόγηση των κατά προτεραιότητα επικίνδυνων ουσιών σε νομοθετικό πλαίσιο. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις πώς θα εφαρμόσετε αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές στην πρακτική. Αφετέρου, εάν όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση δεν αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες κανόνες, εφόσον φυσικά υπάρχουν κανόνες, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα, ότι δεν θα ε, επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις στις ε, επιχειρήσεις πώς αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα πιο επικίνδυνα μείγματα τα οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε πρώτα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα ερωτήσεων μου. Οι δεύτερε ερωτήσει μου, η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων μου αφορά τα επίγοντα ζητήματα. Στο τέλο της ομιλία σα αναφέρατε ότι προβλέπετε να λάβετε κάποια μέτρα άμεσα θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ακριβείς. Τι θα γίνει κατ' επίγον, με, με επίγουσες διαδικασίες και όπως είπε η συναδελφός μου έχουμε ήδη πολλά στοιχεία σε ορισμένες, ε, για ορισμένες περιπτώσεις. Η έκθεση για την τοξικότητα των μειγμάτων έδειξε ότι ορισμένα μείγματα, δηλαδή πολύ περιορισμένο αριθμό προϊόντων είχαν ε, επιβλαβεί συνέπειες. Μήπως θα μπορούσαμε για αυτή την ομάδα προϊόντων, τη μικρή ομάδα προϊόντων, να λάβουμε συγκεκριμένες δράσεις ώστε ακριβώς να ε, περιορίσουμε την έκθεση και τις συνέπειες αυτής της έκθεσης για την δημοσιογεία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μελετάμε τις μεθόδους αξιολόγησης, αλλά πιστεύω ότι για το συμφέρον των συμπολιτών μας το σημαντικότερο είναι να δράσουμε ε, ρεαλιστικά και να ε, αντιληφθούν οι συμπολίτε μας ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για ένα ζήτημα το οποίο επιδεινώνεται σε πολλές χώρες στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το 1999 βρισκόσασταν εδώ. Θυμάστε εκείνη την ανακοίνωση για τους διαταράκτες ενδοκρινικούς. Τι γίνεται. Φανταστείτε. Τα λέγαμε τότε, λέμε και τώρα, έχει την έκθεση κυρία Βέσλη. Φανταστείτε άλλα 13 χρόνια να περάσουν και ακόμα να λέμε τα ίδια, χωρίς να έχουμε καταλήξει σε κάποιο είδου συγκεκριμένο νομοθέτημα. Γι' αυτό σας λέω, με ανησυχεί κάπως αυτή σας η, η προσέγγιση ότι θέλετε πάντοτε να κάτι να έχει έτσι στέρεα θεμέλια, να είναι αδιαμφισβήτητο, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πριν κινηθείτε για οποιοδήποτε είδους ε, θέσπιση νομοθετήματος. Γιατί, τι να σας πω, όταν λέτε επιστήμη, τι επιστήμη στο μυαλό σας. Να, λέω εδώ πέρα, έχει αυτή την έκθεση του Πανεπιστήμιου του, του Γκέτεμπορ, και ό,τι βλέπω δηλαδή για την, για την οικοτοξικότητα, τα αποτελέσματα ε, αυτά δεν σωρεύονται πάντα δεν, δεν μπορούν να θεριστούν και πολλές φορές υπάρχουν υπάρχει ακόμα και συνέργεια στις συνέπειες αυτών των φαινομένων επομένως θέλουμε όσο γίνεται να, είναι στεγανά πλευρά ασφαλεία στις ρυθμίσει αλλά και προηγουμένως του είπαμε ότι αν έχουμε συνδυασμό συγκεκριμένων χημικών ουσιών δεν λέει αυτό τίποτα μπορεί μετά τις κάποιες δοκιμές να αποδειχθεί ότι δεν χρειάστηκε να ήταν τόσο ψηλό το επίπεδο ασφαλείας. Μπορούν λοιπόν να ανακατευθούν αυτές οι ουσίες. Άρα για να αντιστρέψουμε το βάρος της αποδείξεως όπως γίνεται ας πούμε στο Ρίτσο. Εγώ δεν επικρίνω την ανακοίνωση γιατί φυσικά και υπάρχει χρήσιμα στοιχεία. Αλλά αυτό το οποίο θέλω είναι να αναλαμβάνεται δράση κατά συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θέλω να περάσουν άλλα 13 χρόνια. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω για να προστατεύσουμε την ε, την υγεία μας. Δυστυχώς, αυτή η μελετή Επιτροπή δεν χρησιμοποιήθηκε δεν, σε όλες τις διαστάσεις. Και νομίζω ότι το Σκανδιναβικό Συμβούλιο έχει κάποια στοιχεία να συνεισφέρει θετικά. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απάντησή της. Σύμφωνα με την ότι εδώ θα πρέπει να ακολουθούμε την αρχή της σύνεσης. Έχουμε τώρα αυτή την ε, μελέτη που έγινε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω όμως εδώ πέρα ότι χάνεται το δάσου για το δέντρο. Γιατί μιλούμε τώρα για κάποιες συγκεκριμένες ουσίες, λίγες. Τι λέτε. Ακούσαμε για τη συνδυασμένη επίδραση τη συνδυασμένη χρήση χημικών. Θα πρέπει να είναι σαφέστερη η Επιτροπή για το ότι ίσως υπάρχουν αποτελέσματα συνδυασμένης χρήσης. Να δούμε το πώς δρούν αυτές οι χημικές ουσίες επί των ε, αγρίων ζώων και επιδρούν τελικά στα οικοσυστήματα. Αλλά βέβαια και για την ανθρώπινη υγεία. Άρα θα πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα το θέμα και σχέση με την άγρια ζωή και σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Κάπως θα πρέπει να συνδυάσετε, να συντονίσετε την ομοθεσία; Και μετά να προχωρήσετε κάποια ευέλικτη νομοθεσία. Και άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνετε με αυτό το στην ήπια νομοθεσία. Ο Πρόεδρος. Ποιος άλλος θέλει το λόγο τώρα, η Επιτροπή. Για να απαντήσει σε ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις. και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που μου δίνεται η ευκαιρία να σας διαφωτίσω και να προβληματιστούμε λίγο περισσότερο προβληματισμούς που δεν καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στις περιορισμένες σελίδες της ανακοίνωσης για πολλά ζητήματα. Το ζήτημα της αρχής προφύλαξης το υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε αυτή την αρχή και την εφαρμόζουμε όταν είναι απαραίτητο και δυνατό. Και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω γιατί πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπουν την, χωρίς εξαιρέσει την κατηγορηματική εφαρμογή της αρχής προφύλαξης. Αντιθέτως χρειάζεται περαιτέρω εμπειρία και περαιτέρω διερεύνηση. Αλλά ας περάσω πρώτα στις πιο εύκολη ερωτήσεις όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας. Πώς θεωρούμε ότι θα εργάζεται αυτή η ομάδα εργασίας. Έχουμε καλέσει μια πρώτη συνάντηση των σχετικών ενδιαφέρομενων οργανισμών και αρχών και των υπηρεσιών της Κομισιόν ώστε να συζητήσουμε ακριβώς πώς θα πρέπει να συνεργαστούμε και πώς θα εφαρμοσουμε τη διαφάνεια προς τους έξω εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους από τις πράσινες μη κυβερνικές οργανώσεις, τους οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών και τις βιομηχανίες. Δεν το συμπεριλάβαμε στην ίδια ανακοίνωση αυτό, διότι θεωρήσαμε ότι αυτό το ζήτημα χρειάζεται λεπτομερή συζήτηση. Αυτό όχι διότι δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς, αλλά διότι το θέμα είναι σύνθετο. Και το να έχουμε πολλούς ανθρώπους μέσα σε μια αίθουσα που να συζητάνε για ένα δύσκολο θέμα είναι κάτι δύσκολο. Θα συναντηθούμε λοιπόν εντό τη Κομισιόν με τους συναδέλφους μα, ώστε να, δούμε, να βρούμε τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης αυτής της συνεργασίας. Αλλά ευχαρίστω σα σας αναφέρουμε σε τακτικά διαστήματα εφόσον θέλετε σε αυτή την Επιτροπή για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί και ειδικότερα θα σας ε, κάνουμε μια έκθεση εγγράφου στο, έως το 2015, αυτό είναι σαφές. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει βούληση για να είμαστε ανοιχτοί και να εμπλέξουμε και άλλους ενδιαφερομένους, αλλά κοίταμε να δούμε τις πρακτικές λεπτομέρειες. Για να πω τώρα στις πιο δύσκολες ερωτήσεις και να προσπαθήσω να δώσω μια ικανοποιητική απάντηση. Θα πλησιώσω κάπως στην απάντησή μου με την πρόταση για το Συμβούλιο των Βόρειων Χωρών και τη χρήση της αρχής της προφύλαξης λέγοντας ότι ήταν σαφές ε, από την έκθεση που αναφέρατε, Κορτεν Κάμπ, και ε, από τη γνωμοδότηση που λάβαμε από τις επιστημονικές επιτροπές ότι ελάχιστη νομοθεσία ισχύει σήμερα που να καλύπτει τα τυχαία μείγματα. Έχουμε ισχύουσα νομοθεσία για πολύ συγκεκριμένα μείγματα τα οποία δημιουργούνται εσκεμένα. Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, είναι τα πιο χαρακτηριστικά και πιο γνωστά. Αλλά ελάχιστη νομοθεσία μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τυχαία μείγματα. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα έχει κάποιους κανόνες που μας το επιτρέπουν, αλλά σίγουρα στο βαθμό που αναφέρεται ως επιθυμητός ε, στην έκθεση και στην επισκόπηση της, ε, στην αναθεώρηση της, των επιστημονικών επιτροπών. Έχουμε λοιπόν σποραδική νομοθεσία που καλύπτει πολύ συγκεκριμένα μείγματα, αλλά σίγουρα όχι ολόκληρο το εύρος ε, πιθανών μειγμάτων. Η συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας γίνεται με δύο τρόπους. Ε, ο πρώτος είναι ότι όλοι οι επιστήμονες που συμβουλευτήκαμε, όπως και ο καθηγητής ε, Κόρτεν Κάμπς και η ομάδα που το βοήθησε για τη σύνταξη της έκθεσής του, της μας είπαν ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά μείγματα στα οποία είναι εκτεθειμένοι οι άνθρωποι και το περιβάλλον αλλά ότι είναι πολύ πιθανό, ότι πιθανότατα ο η πλειοψηφία αυτών δεν είναι ανησυχητική. Από την άλλη έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπως επισημάνθηκαν στην έκθεση Cotton Κάμπ, όπου υπάρχει έκθεση σε μείγματα ανησυχητικά. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα δεδομένων των σημερινών ωστόσο επιστημονικών στοιχείων που μας έχουν παρασχεθεί, ειδικότερα μέσω των επιστημονικών επιτροπών, είναι δύσκολο να κρίνουμε την έκταση του προβλήματος. Να εκτιμήσουμε την έκταση του προβλήματος ειδικότερα διότι συνεννούν όλοι οι επιστήμονες ότι πολλά από αυτά τα μείγματα δεν είναι ανησυχητικά. Υπάρχει λοιπόν μια γκρίζα ζώνη στο ενδιάμεσο όπου θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την έκταση του προβλήματος και αυτό αποτελεί κίνητρο για τη συστηματική εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης ε, μέσω της ε, ανακοίνωσης της Κομισιόν να γνωρίσουμε καλύτερα την έκταση του προβλήματος. Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά σε μια ερωτήσεις, ε, έχουμε από την Επιστημονική Επιτροπή μας λένε ότι πιστεύουν ότι τα μείγματα συμπεριφέρονται διαφορετικά. Έχουν διαφορετική τοξική επίδραση στο περιβάλλον από τον στον άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα στην προσέγγιση μας. Μας λένε οι επιστημονικές επιτροπές ότι οι συνδυασμένες επιδράσεις συγκεκριμένων συγκεντρώσεων στο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα και ε, κατά πόσο αναθριστούν αυτές οι συγκεντρώσεις ε, είπαν οι επιστημονικές επιτροπές ότι για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να υπάρχει τέτοια συνάθρηση εφόσον ε, η έκθεση σε ένα επιμέρους ε, συστατικό είναι χαμηλότερη από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τότε δεν χρειάζεται να φοβόμαστε συσσόρευση των επιδράσεων. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία, πρέπει να τα μελετήσουμε, να τα κατανοήσουμε ω Κομισιόν στην ομάδα εργασία. Απ' την άλλη, είναι δύσκολο να καταλάβουμε την εκτέλεση του πρόβληματο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι έτσι όπω έχουν τα πράγματα και αντίθετα από ό,τι συνέβη με την ανακοίνωση του 99 για του ενδοκρινικούς διαταράκτε, δεν μπορούμε απλά να εκδώσουμε μία σύσταση για να συμπληρώσουμε τα κενά που έχουμε στη γνώση μας πρέπει να λάβουμε και συγκεκριμένες δράσεις. Συγγνώμη, αυτό αναφέρονταν στην ανακοίνωση του 99. Υπάρχουν δύο δράσεις ουσιώδους περιεχομένου που δεν εντάσσονται στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Θα εξετάσουμε μείγματα, υπάρχουν τα μείγματα και ειδικότερα θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία αυτά που αναγνωρίζει ο καθηγητής Κόρτεν Κάμπ στην εκθέσή του καθώς και εκείνα που εντοπίστηκαν από τις επιστημονικές επιτροπές στην αναθεώρηση της έκθεσης ώστε να κάνουμε μελέτες πραγματικών περιπτώσεων. Και έτσι γίνεται σαφές ε, ε, ότι αυτό, ε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη προσέγγιση χωρίς αβεβαιότητες και φυσικά δεν μπορούμε ακόμα να προσδιορίσουμε ακριβώς το πρόβλημα, αλλά η οι δυσκολία στον έλεγχο τη έκθεση σε μείγματα δεν αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητα, διότι ο καθηγητή Κόρτεν Κάπ με τη βοήθεια τη Επιστημονική Επιτροπή ε, μας παρήχε τεχνικές για να το πράξουμε αυτό. Ο δύσκολο, οι μεγάλε προκλήσει είναι στην εκτίμηση της αντιμετώπισης, διότι πρέπει να επιλέξουμε το συστατικό του μείγματος, που είναι αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε πιο στεναρά από τα υπόλοιπα. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατά, κατά περίπτωση προσέγγιση, όπως αναφέρουμε στην ανακοίνωση, βάσει εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά. Τέλος, ε, όσον αφορά την καθοδήγηση, Σκοπός ε, δεν είναι εδώ να είναι αυτή η κυρία δράση. Σκοπός είναι ότι θέλουμε να αναπτυχθεί η καθοδήγηση ειδικότερα σε δύο τομείς. Στο πρόγραμμα για τα φυτοφάρμακα η ΕΦΣΑ αναπτύσσει καθοδήγηση όσον αφορά την τοξικότητα μειγμάτων για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, χημικών που δρούν με τον ίδιο τρόπο και στο κανονισμό των βιοκτώνων ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών θα πρέπει να κάνει κάτι παρόμοιο αλλά λίγο πιο ευρέως. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι η καθοδήγηση, οι κατευθυντήρε γραμμέ, ειδικά εκεί, θα πρεπει να κανει κατι παρομοιο αλλα λιγο πιο ευρεως και αυτο που θελουμε να κανουμε ειναι να διασφαλισουμε οτι η οι κατευθυντηρε γραμμε ειδικα εκει θα βασιστουν σε παρόμοιε έννοιε, αλλά και ότι αυτέ οι δύο καθοδηγήσει θα μα οδηγήσουν σε μια, σε γραμμή που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε νομοθετικό ε, πλαίσιο σε περίπτωση που χρειάζεται αυτό το νομοθετικό πλαίσιο να αξιολογήσει ένα μείγμα. Αλλά θέλω να επισημάνω αυτό που θεωρούμε σημαντικό κίνητρο για δράση στην ανακοίνωση πέραν των σαφώ αναγκαίων δράσεων για την κάλυψη των κενών γνώσεων στην παρακολούθηση και την τοξικότητα που είναι ουσιαστικέ δράσει, είναι η δράση του να πάρουμε πραγματικά μείγματα για τα οποία έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο αυτών και να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί η διαχείριση επικίνδυνότητα για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Um, Δεν ήθελα να είμαι κάστορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μερικές ακόμη ερωτήσεις. Όταν παραδεχτήκατε ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τις επιδράσεις αυτών των χημικών, είμαι βέβαιος ότι θα πάτε πίσω στην Κομισιόν, στον αρμόδιο επίτροπο για το ορίζοντα 2020 και θα τον ενημερώσετε για αυτές τις ανάγκες για μεγαλύτερη γνώση και έρευνα σε αυτό το τομέα με τα επίσης όταν διοργανώσετε το συνέδριο και καλέσατε κόσμο για να συζητήσετε αυτό το πρόβλημα παρακαλώ μην επαναλάβετε το τόσο συχνό λάθο, σε τόσους πολλούς φακέλους ε, όπου οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας κατέχουν το 80% των θέσεων ε, στην αίθουσα να συμπεριλάβετε ένα τρίτο και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερομένους να υπάρχει μια ισορροπημένη συζήτηση ένα ισορροπημένο κοινό που συζητάει και όπως γνωρίζετε εγώ είμαι χημικός. Μία από τις εμπειρίες μου στο πανεπιστήμιο ήταν ότι κάναμε κάποια πειράματα και συνήθως τα απολύματα τα χύναμε στον νεροχύτη και μια μέρα ξαφνικά είδαμε ένα σύννεφο, ένα νέφος καπνού που άρχισε να ενοχλεί τους ε, συναδέλφους μου και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι συνέβη μέσα σε αυτόν τον νεροχύτη και με τη βοήθεια του καθηγητή μας καταλάβαμε ότι δημιουργήσαμε ένα πραγματικά τοξικό, σοβαρά τοξικό συστατικό με μη τοξικά συστατικά που ρίξαμε στο νεροχύτη. Τότε δεν το αντιληφθήκαμε όταν ρίχναμε αυτά τα συστατικά στο νεροχύτη, αλλά όταν το μελετήσαμε και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι συνέβη μέσα σε αυτό το νεροχύτη, αντιληφθήκαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα τυχαίο μείγμα Μπορεί ένα μείγμα να είναι τυχαίο, αλλά μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί όταν, ας πούμε, ρίχνεται στο νεροχύτη της κουζίνας, ε, χρησιμοποιείται, ας πούμε, χλωρίνη για να καθαρίσετε τις ολίνες ή διάφορα καθαριστικά. Μπορεί να δημιουργηθούν τυχαία μείγματα, τα οποία βεβαίως ε, εύλογα μπορούν να προβλεφθούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να τα προβλέπουμε και να αναλαμβάνουμε δράση. Τώρα είναι δύσκολο να θυρωθεί ένα ασφαλές επίπεδο έκθεσης ήδη για ένα υπάρχουν χημικό, πόσο μάλλον για μείγματα χημικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια αρχή προφύλαξης, διότι η επιστήμη για την καθιέρωση ενός ασφαλούς επίπεδου για όλα αυτά θα μπορούσε να καταναλώσει όλο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια μέθοδο προφύλαξη ε, για την προσέγγιση όλων αυτών, διότι διαφορετικά θα ξέψουμε όλα μα τα λεφτά προσπαθώντα να ορίσουμε αυτά τα επίπεδα. Χρειαζόμαστε κάποια λογική προσέγγιση. Θέλετε να απαντήσετε και σε αυτό. Μου επιτρέπετε. Πολύ ευχαριστώ. Θα απαντήσω. σα ευχαριστώ θερμά. Μια εξισορροπημένη προσέγγιση. Βεβαίως και συμφωνώ ότι υπάρχει τέτοια ισορροπημένη, σταθμισμένη προσέγγιση και αυτό έχει κάνει και η Επιτροπή. Τότε που συγκροτήσαμε αυτές τις ομάδες των ειδικών για να εξασφαλίσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Επομένως, γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους. Σίγουρα και συμφωνούμε με αυτό. Οπότε βέβαια ο μηχανισμός του να γίνει αυτό, το πώς θα γίνει δηλαδή, αυτό εντάξει θα πρέπει να το βρούμε. Τόσο αφορά τα ατυχήματα στο σπίτι. Υπάρχει πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει δηλαδή όσον αφορά τον κανονισμό για την ε, γεωτοδεσία, τη, τη συσκευασία, την κατηγοριοποίηση και λέω ότι έτσι θα πρέπει να ενημερώσουμε αυτέ τι ε, πληροφορίε σε σχέση με τα κέντρα δηλητήρια στα εθνικά και το ατύχημα εάν οδηγεί σε πρόγραμμα, σε πρόβλημα συγγνώμη, υγείας, ε, ζαλάδες, αυτοί σε κάτι τέτοιο, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στο κέντρο δηλητηρίας. Και έτσι να έχουμε ένα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τουλάχιστον Έτσι τουλάχιστον ξέρουμε τι γίνεται για να αντιδράσουμε. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουμε. Ε, αυτό απομένει να μελετηθεί σε σχέση με τον κανονισμό αυτών που τον προϋπάρξει, το είπαμε για την κατηγοριοποίηση, κατάταξη, ξέρω εγώ, ταξινόμηση ή αλλιώ. Τώρα, όσον αφορά τα επίπεδα ασφαλεία, καταλαβαίνω, ξέρω από πού προέρχεστε, που το πάτε, τέλος πάντων, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε σήμερα είναι ότι το ΡΙΤΣ έχει ορίσει κάποια όρια ασφαλείας για κάθε χημική ουσία, όμως υπάρχει αυτό το όριο των δεκατών καινούριο. Και επομένως έτσι υπάρχουν κάποια τέτοια όρια. Και ρυθμίζεις μετά για κάθε χημική ουσία. Οπότε άπρος και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες για το κάθε χημική ουσία, που θα μπορούμε να καθορίσουμε με με τεχνικές όπως την έκθεση Κόρτεμπαχ σε σχέση με το μείγμα οπότε ίσως θεωρείται ότι δεν αντιδράσαμε ταχύως αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια μελέτη αναπερίπτωση δυνάμει των όσων επιτάσσει ο κανονισμός του Ρίτσου σίγουρα με πληροφορίε. Υποχρεώνουμε τη βιομηχανία να μα στέλνει πληροφορίε. Έτσι βελτιώνουμε τη γνώση μας. Και καταλήγουμε μετά στη συγκεκριμένα μείγματα στο τι θα ίσχυε. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Και όλους τους συνοδέλφους που λαμβανούν μέρος στη συζήτηση. Πέρα στη συνεδρίαση σήμερα. Αύριο στις 10 το πρωί. Θα έχουμε τον κύριο Στόιμπερ. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε ασφαλώς. Γιατί πρόκειται για του ανεξάρτητου ενδιαφερόμενου φορεί και την ομάδα υψηλού επίπεδου για το διοικητικό φόρτο. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο το πρωί. Καλό σα βράδυ.